καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία των Πεσμεργά από το αυτόνομο Κουρδιστάν του Ιράκ υπό την ηγεσία ε, του στρατηγού Τζαφάρ Αλή. Είναι ένοπλα τμήματα των Κούρδων στο Ιράκ, στο θεωρείο των επισήμων.